της συνεδριάσεως δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι ε, είμαστε πάλι σε απευθείας μετάδοση από το διαδίκτυο, σε web stream. Αυτά δηλαδή τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα μπορεί να τα παρακολουθήσει ο καθής από ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου και αισθανόμαστε ιδιαίτερη περηφάνεια για αυτή τη δυνατότητα τη τεχνολογία. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε από το να εγκρίνουμε την έκθεσή μα και να ψηφίσουμε τι τροπολογίε. Εάν τυχόν οι δύο ώρες που είχα προβλέψει εγώ τουλάχιστον δεν μας αρκέσουν, μάλλον μας αρκέσουν, δεν θα χρειαστεί να κάνουμε συνεδρίαση αύριο. Φαντάζομαι δεν έχει κάνει αντίρρηση σε αυτό. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι είχαμε στο παρελθόν κάποιες δυσκολίες λόγω ταυτόχρονης διεξαγωγής συνεδριάσεων και ψηφοφοριών σε άλλες επιτροπές. Παρακαλώ όμως να επισημάνουμε ότι οι άλλες επιτροπές που ενδεχομένω έχουν ταυτόχρονα μα ψηφοφορίε, είχαν και άλλες ευκαιρίε και άλλα δηλαδή χρονικά σημεία στα οποία μπορούσαν να προβλέψουν τις ε, ψηφοφορίες του ενώ εμείς μόνο μία επιλογή είχαμε και δει μια επιλογή η οποία είχε προσδιοριστεί από πέρσι το Σεπτέμβριο συγκεκριμένα 25 Μαΐου το απόγευμα από τις 3 και μετά και 26 το πρωί. Εάν κάποιος δεν μπόρεσε να έρθει για να ψηφίσει, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ας κανονίσει ο καθένας την πορεία του. Αυτά. η επιστολή που μου απέστειλε η Ντανούτα Χούμπνερ, πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, όπου μου προτείνει να μην τοποθετηθούμε σε θέματα περιφερειακής πολιτικής τόσο αναλυτικά και στην οποία μου επεσήμενε ότι θεωρεί πως οι τροπολογίες και συμβαστικές τροπολογίες για τις ενδιάμεσες περιφέρειες δεν είναι παραδεκτές. Έλαβε απάντηση από πλευρά μου. Τη απέστειλε λοιπόν και εγώ μια επιστολή όπου τη είπα ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η εντολή μα και η εντολή μα είναι να διατυπώσουμε νομοθετικό έργο. Μπορούμε δηλαδή να απαλλάξουμε από το βαρύ καθήκον της νομοθετικής, νομοθετικού έργου και την Επιτροπή των Περιφερειακών θεμάτων, διότι έχουμε να διατυπώσουμε προτεραιότητες και ιδέες, θέσεις, τοποθετήσεις και για τα δημοσιονομικά θέματα όπως και για τα περιφερειακά. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν θελήσαμε να επεκτείνουμε πολύ αυτό το πεδίο. Απλώς σας το λέω για να ξέρετε τι είδους απάντηση δόθηκε. Μετά τις ανακοινώσεις αυτές και για τελευταία φορά πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Γκαρίγα για την παρουσίαση της έκθεσης του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω τεχνικού τύπου σχόλια. Να σας πω μόνο ότι έχετε 114 συμβαστικές τροπολογίες, συν κάποιες προφορικές, συν μερικές εναλλακτικές τροπολογίες ε, που αποτελούν το επιστέγασμα εργασιών ενός έτους και πολλών συνεδριάσεων της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Προέκυψαν όλα αυτά από πάνω από χίλιες ε, προτάσεις τροπολογιών που κατατέθησαν. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την γραμματεία, ιδιαίτερο την Μόνικα Στράσερα αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό και κατόπιν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δικούς μου βοηθούς, τους συντονιστές των άλλων πολιτικών ομάδων που ε, διαπραγματεύτηκαν μέχρι τελευταία στιγμή κάνοντας τη ζωή μου δύσκολη ε, το κείμενο αυτό. Ελπίζω να τελειώσουμε σε δύο ώρες όπως ακριβώς μας καθοδηγεί η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Σαλβαδόρ, προφανώς και θα συνέβαινε αυτό. Είσαι έμπειρος συνάδελφος, ξέρεις ότι ποτέ δεν έχει ο εισηγητής εύκολο καθήκον, όποια έκθεση και να αναλάβει. Να σας ενημερώσω για κάποια τεχνικά θέματα, αλλά πρώτα να δώσω το λόγο στην Αν ε, Γένσεν. Ίσως πρόκειται για ένα τεχνικό σχόλιο. Στην ομάδα μου εκπλαγήκαμε από το γεγονός ότι οι γνωμοδοτήσεις των υπολείπων επιτροπών είναι στον κατάλογο ψηφοφοριών. Ορισμένες επιτροπές έχουν ψηφίσει, ορισμένες άλλες όχι. Ε, ο εισηγητής έχει σημειώσει με μείον όλες τις προτάσεις. Βέβαια, φοβόμασταν ότι έχοντας αυτές τις νομοδοτήσεις στον κατάλογο ψηφοφορίας, ε, ίσως θα μπορούσαμε να θολώσουμε όλη την έκθεση και να πάψει να είναι έτσι λογικά συνεπής η έκθεση. Ε, εξ αρχής εμείς είχαμε πει ότι η διαδικασία δεν ήταν πολύ σωστή με γνωμοδοτήσεις από διαφορετικές επιτροπές ε, διότι θα έπρεπε οι παρόντες να υποβάλουν τροπολογίες και ε, όχι να λάβουν υπόψη τις τροπολογίες κατευθείαν από τις επιτροπές. Ναι, σαφώς. Από την αρχή είπαμε ότι θα λάβουμε υπόψη οτιδήποτε μας έχουν κοινοποιήσει είτε μέσω επιστολής είτε μέσω ε, μιας πιο τυπικής ε, διαδικασίας ψηφοφορίας ή λοιπές επιτροπές. Ως προς το περιεχόμενο. Αυτό είπα. Τα λαμβάνουμε υπόψη. Και αν δείτε τις συμβαστικές τροπολογίες νομίζω ότι φαίνεται σαφώς πως ε, έχουμε συμπεριλάβει τα θέματα και τις παρατηρήσεις των λοιπόν επιτροπών. Αλλά εγώ επιλογή άλλη δεν έχω, περιθώριο άλλο, από αυτό που μου ορίζει η εντολή μας η οποία λέει στο άρθρο 49 ότι εμείς αποφασίζουμε και ψηφίζουμε την έκθεσή μας. Τελεία και παύλα. Γι' αυτό οι παράγραφες εκείνες οι οποίες... Οι παράγραφοι εκείνες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από τις συμβαστικές τροπολογίες επανέρχονται στον κατάλογο των ψηφοφοριών εμφανίζονται δηλαδή και πάλι και αν συμφωνούν οι συνάδελφοι μπορούμε για να επιταχύνουμε τη διαδικασία να πούμε ότι εάν υπάρχουν περισσότερες από τις τροπολογίες μίας ε, συγκεκριμένης επιτροπής μπορούμε να τις εγκρίνουμε, να τις ψηφίσουμε όλες μαζί on ε, block αλλά τίποτε περισσότερο από αυτό που λέει ο κατάλογος ψηφοφοριών δεν μπορώ να κάνω. Πριν τώρα περάσω στην ανακοίνωση των λοιπόν τεχνικών θεμάτων, θα πρέπει να πω κάτι που χαλισμονεί στην αρχή. Να υπενθυμίσω ότι πρέπει κανείς ε, ο κάθε ένα από τους συναδέλφου που έχουν το δικαίωμα συμμετοχή στην ψηφοφορία να ελέγξει αν έχει την κάρτα του μαζί. Την κάρτα για τις ψηφοφορίες. Δεν βλέπω να αναπηδά κανεί και να λέει Παναγία μου, Παναγία μου το ξέχασα. Άρα μάλλον καλά, καλό δείγμα είναι αυτό. Αλλά ας κάνουμε μια επαλήθευση της, ε, των τεχνολογικών των τεχνικών εγκαταστάσεων. Μια πρώτη δοκιμή λοιπόν, ψηφοφορία, Φερρυπίν. Η Επιτροπή Σούρε έκανε καλή δουλειά. Ναι, ου, αποχές. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγώ δεν, δεν συμμετέχω στην ψηφοφορία, λέει η Πρόεδρος. Die... Die τη ψηφοφορία. Αυτό και είναι καλό αποτέλεσμα. 51 εψήφισαν. 40, μάλλον είχαν δικαίωμα ψηφοφορίε. 48 εψήφισαν. 33 θεώρησαν ότι ήταν καλό το αποτέλεσμα. Ένας ε, ψήφισε αρνητικά και οι υπόλοιποι 14 δεν ήταν και πολύ σίγουροι. Εν πάση περιπτώσει όμως είδαμε ότι τουλάχιστον δουλεύει το σύστημα. Εψήφισαν 51. 50 όμως είναι τα μέλη της Επιτροπής. Ας επαληθεύσουμε λοιπόν από ποια ομάδα είναι περισσεύει κάποια ψήφος. Ah ja, okay. Trotzdem nur, Ah, okay, okay, alles klar. Okay, gut, gut, gut. So. Also, ein Elliot, genau. Das ist der gute Geist. Ναι, ναι. Το καλό πνεύμα της Ανέλιωτ είναι μαζί μας μεχρικά τεχνικά ζητήματα ακόμα. Υπάρχουν στη διάθεσή σας σε κάθε γλώσσα οι τροπολογίες στο σύνολό τους, πιστεύω να το έχετε δει όλοι. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες, όπως είχαμε συμφωνήσει, είναι διαθέσιμες στα αγγλικά στο σύνολό τους. Ο κατάλογος των ψηφοφοριών έχει αποσταλεί σε όλους τους αδέλφους και στις ομάδες ώστε να μπορέσουν και οι ομάδες να κάνουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους ως προς που θα τηρήσουν σε κάποιες ψηφοφορίες για τροπολογίες. Στις συμβιβαστικές τροπολογίες όταν υπάρχουν, σαφές είναι ότι οι συμβιβασμοί που έχει προτείνει ο ίδιος ο εισηγητής είναι αυτοί που ψηφίζονται πρώτοι. Εάν ζητήσει κανεί κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να το απορρίψω. Αυτό ορίζει ο κανονισμό στην παράγραφο 160. Επομένω. Μάλλον 61, συγγνώμη. Επομένω, πρώτα ψηφίζεται η συμβαστική τροπολογία του εισηγητή. Στη συνέχεια βλέπουμε αν υπάρχουν κάποιες άλλες τροπολογίες οι οποίες ενδεχομένω έχουν καλυφθεί και επί... εκ τούτου καταπίπτουν από την συμβαστική τροπολογία και έτσι προχωρούμε. Υπάρχουν κάποιε προτάσει επίση, στι οποίε ε, ζητείται η συμπλήρωση κάποια τροπολογία με μέρο κειμένου. Όπου συμβαίνει αυτό, επιτρέπεται φυσικά, το επισημαίνει ο κατάλογος των ψηφοφοριών. Δεν υπάρχει κίνδυνος δηλαδή για τέτοιου είδου ε, προβλήματα υπαρξή. Έχω δύο αιτήματα λάβει για προφορικές τροπολογίες. οι οποίες όταν έρθει η σειρά τους θα αναγνωστούν, ε, αλλά εάν κοιτάξετε στο τέλος του καταλόγου των ψηφοφοριών τις έχουμε συμπεριλάβει τις προφορικές τροπολογίες έτσι ώστε να μην είναι μόνο προφορικές αλλά να μπορείτε να τις λέτε και γραπτά. Αυτά. Ελπίζω να τα κάλυψα όλα. και να μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Παρακαλώ, πάρτε στα χέρια όλοι τον κατάλογο των ψηφοφοριών ή αν δεν σας ενδιαφέρει αφήστε το πάνω στραπέζι σας και ξεκινάω με την ψηφοφορία για τον τίτλο. Υπαριθμόν ένα τροπολογία τίτλος εκθέσεως. αν θέλετε και διανατάσσεως μπορούμε να ψηφίσουμε, υπέρ της τροπολογίας παριθμών 1. Κατά. Η πλειοψηφία κατά... Αποχές. Ελέγξτε, λένε οι πράσινοι. Καλώς. Άρα προχωρώ στο πρώτο τμήμα. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 4. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. Υπαριθμόν 5 τροπολογία. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Τρεις ψήφοι κατά, δύο αποχές εγκρίνεται. Συμπλήρωση στο κείμενο της ε, παραγράφου 2 με την τροπολογία 80 παρακαλώ υπέρ κατά δεν βλέπω να σηκώνει κανείς το χέρι του στο υπέρ άποχες Ούδης. Απορρίπτεται. Αλλάζω σελίδα, πάω στο δεύτερο. Τροπολογία υπαριθμών 86. Υπέρ. Αυτό. Κατά. Περισσότερο από 8. Αποχές. Ούδης. Τροπολογία παριθμών 87 υπέρ. Αρκετή, αρκετή, αρκετή, αρκετή. Περισσότερη. Ας κάνουμε ηλεκτρονικά την ψηφοφορία απευθείας για να μην χάνουμε χρόνο. Παρακαλώ, ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Die S&D hat ein zu viel. Οι σοσιαλιστές έχουν έναν ε, Εγώ δεν ψήφισα καν, λέει ο πρόεδρος. Καλώς, βγαίνει ένας λοιπόν. «24 υπέρ, 23 κατά, μία αποχή εγκρίνεται». Kommen wir zu 88. Στην τροπολογία 88 τώρα. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Πέραση τη ψηφοφορίας. Οι CNR έχουν έναν ε, παραπάνω βουλευτή. Πέρα τη ψηφοφορία. 23 υπέρ. 22 κατά. Δύο εποχές. Στενές Θα δούμε αν χρειαστεί να ξανακάνουμε ηλεκτρονικά. Συνεχίζουμε με την 89 ηλεκτρονικά για να μην χάνουμε χρόνο. Πέρας. 14 υπέρ, 31 κατά, 2 αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Ουδής. Αποχές. Ουδής. Ομόφωνα λοιπόν εγκρίνεται. Στην 99. 99. Ε, καλύπτεται από την συμβαστική 9. Εάν εγκρίνουμε τι συμβαστικέ 9 και 34, καλύπτεται η 99, αλλά αυτή τη χρονική στιγμή δεν γνωρίζουμε αν θα καλυφθεί και άρα πρέπει να την ψηφίσουμε. 99. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Καλώς. Συμβαστική 7. Κατά. Αποχές, αποχές ομόφωνα λοιπόν εγκρίνεται, δεν υπάρχουν ούτε αποχές στο ψήφι Και προχωρώ στην 105, υπαριθμόν 105 τροπολογία υπέρ. Κατά. Η πλειονότητα από ό,τι φαίνεται, αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Ουδής, αποχές. Ουδής, ομόφωνα εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέρ. κατά ουδείς αποχές α, μία αποχή μία αποχή λοιπόν και κατά τα άλλα εγκρίνεται από όλους τους άλλους και τώρα πρέπει να σφίσουμε τροπολογία υπαριθμών 111 για την παράγραφο 5 υπέρ της τροπολογίας 111 2 κατά περισσότεροι από δύο αποχές Απορρίπτεται. 113. Κατά. Αποχές. Ουδής. Απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία. 112. Υπέρ. Κατά. Περισσότεροι από έξι. Αποχές. Απορρίπτεται. 114. Δεν ξέρω αν φαίνεται τόσο ξεκάθαρα. Κατά παρακαλώ. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. 114 ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. 18 υπέρ. 28 κατά. Δεν είναι τόσο στενά τα αποτελέσματα, αλλά από εδώ πάνω που κάθομαι δεν φαίνεται τόσο καλά. 115. Έξι. Κατά Περισσότεροι από 6. Αποχές. 2. Απορρίπτεται. 116. 2. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117. 2. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 118. 2, 3. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. 6 κατά. Περισσότερο από έξι. Αποχές. Απορρίπτεται. Επιτροπή Γυναικών τώρα. Τροπολογίε παριθμών 1 και 2 τη Επιτροπή Γυναικών. Μπορούμε να τι ψηφίσουμε μαζί. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Όχι. Όχι. Υπαριθμών 1 τη Επιτροπή Γυναικών. Υπέρ. Κατά. Περισσότερο από 6 αποχές ουδής απορρίπτεται Επιτροπή Γυναικών 2 Επιτροπή Υπερθμών 2 της Επιτροπής Γυναικών 2 υπέρ κατά παρακαλώ Περισσότερο από 2 αποχές απορρίπτεται η τροπολογία Περιθμών 120 τώρα υπέρ 2 κατά περισσότερο υπό 2 Αποχές. Ουδής. Απορρίπτεται. 121. Υπέρ. Έξι. Κατά. Περισσότερο. Αποχές. 122. υπέρ. 6 πάλι. Κατά. Περισσότερο από 6. Αποχές. 123. Άρα ταυτόσιμη, συγχωρείτε, 124. 2 Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126. 2. Κατά. Όλοι οι λοιποί, αποχές, απορρίπτεται. 127. Δύο πάντα. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική παριθμόν 10 υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Κανείς εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβαστική 11. Κατά. 5. 5 ψήφοι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 139. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. 139. Πέρασε φορέας. 19 υπέρ, 29. Γιατί δεν βλέπουμε τόσο καλά την τάση ε, ε, εκ των υστέρων. Πρέπει να σας πω ότι θαυμάζω τους ε, προέδρους ε, στην Ολομέλεια που μπορούν να παρακολουθήσουν την τάση της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 29 κατά. 140. Το ίδιο είναι, η ίδια αναλογία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. 25 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. Υπαριθμόν 12 συμβαστική υπέρ. Κατά. Τέσσερις. Αποχές. Εγκρίνεται. Μάλιστα. Τώρα ξαναρχίζουμε την ουσία στις ψηφοφορίες. 151 παρακαλώ, υπέρ. Ένας κατά. Περισσότεροι αποχές. Απορρίπτεται. 152. Δύο. Ε, κατά παρακαλώ. Περισσότεροι αποχές. Απορρίπτεται 153 υπέρ. 6. Κατά. Περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. 154. Κατά παρακαλώ. Μάλιστα η πλειοψηφία. Αποχές Απορρίπτεται 155 υπέρ. 3 κατά. Περισσότερο. Αποχές. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Ας επαληθεύσουμε. Πέραση στις 23 υπέρ, 24 κατά, μία αποχή, απορρίπτεται. 157 υπέρ. Το ίδιο. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 19 κατά, ουδεμία αποχή, εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Περισσότεροι από 6. Αποχές. Απορρίπτωτη. 160 υπέρ. 7, 8, 9, κατά. Περισσότεροι από 9 αποχές. Απορρίπτεται. 161. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162. Παρακαλώ, James Ellis. Αποσύρω. Η 165 ήταν η δική σου, από ό,τι ξέρω. Ναι, Πρόεδρε, και την αποσύρω. Και σας ενημέρωσα πριν από την αντιεξαγωγή της ψηφοφορίας. 162. Υπέρ. 3. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 165 όπως ακούσατε έχει αποσυρθεί. Τροπολογία συμβιβαστική υπαριθμών 13. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 167 Ένας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. 173. Κατά. Περισσότερο. Κύριε Κοτμάνης. Απορρίπτεται. 172. Κατά. Περισσότερο. Αποχές. Ουδεμία απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπερφών 14 υπέρ. Κατά. Ουδής κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 16 συμβαστική τροπολογία υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Την 8 και 9 μπορούμε μαζί, το περιβάλλοντος, της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Όχι. Καλώς. Υπαριθμόν 8 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Υπέρ. 7. Κατά. Περισσότερες από 7 ψήφοι. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. 2. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ υπάρχει πρόβλημα στη μετάφραση στο αγγλικό κείμενο, ε, στην διερμηνία. Έχω ανοιχτό το μικρόφωνο, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω. Συμβαστική 18. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 197 ως προσθήκη. Ως προσθήκη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Kommt Closed. 25 dafür, 20 dagegen, eine Enthaltung angenommen. 25 υπέρ, 20 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. 201 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή, μία ψήφος κατά. Ακόμα δεν έχετε διερμηνία. Φαίνεται ότι ένα μικρόφωνο δεν δουλεύει στην... ή τα μικρόφωνα δεν δουλεύουν στην αγγλική καμπίνα. Απορρίπτεται. Ε, ακούγεται τώρα η αγγλική καμπίνα. Ακούτε τώρα την αγγλική διερμηνία. Κανονικά ναι, πρέπει να ακούγεται. Πρέπει να ακούγεται τώρα. Ένταξη. 202 στα γερμανικά. Υπέρ της 202 παρακαλώ. Τέσσερις βλέπω. Κατά. Περισσότεροι από τέσσερις. Μάλλον θα πρέπει να πάω στο κομμωτήριο αφού είναι haircut. Ράιμαρ. 205. Δύο. Κατά. Περισσότεροι από δύο εποχές. Ουδής απορρίπτεται. 206 υπέρ... Συγγνώμη, υπέρ, υπέρ. 206, ποτέ δεν είναι κανείς υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Ομόφωνα κατά. Απορρίπτεται. Υπαριθμόν 19 συμβιβαστική παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Τέσσερις. Τέσσερις κατά αποχή, αποχές. Ουδής εγκρίνεται. Γυρίζουμε σελίδα. Η τροπολογία 214. 214 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία ψήφος κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται συμβαστική 21. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές με μία ψήφο κατά εγκρίνεται η τροπολογία 231 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία συμβιβαστική 23 υπέρ κατά τέσσερις αποχές απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη, λέει Πρόεδρος. 230 5.235, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Ουδής. Εγκρίνεται. Επιτροπή Βιομηχανίας Περιθμών 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 245, τροπολογία 245 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 246 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 247. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Με ολίγες ψήφους κατά εγκρίνεται 252 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 12 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ 6 κατά η υπόλοιπη απορρίπτεται ε, αποχές συγγνώμη λέει πρόεδρος απορρίπτεται συμβαστική 26 υπέρ κατά μία ψήφος αποχές ουδής εγκρίνεται 256 256 τροπολογία υπέρ παρακαλώ 4 κατά οι υπόλοιποι αποχές ουδής 257 υπέρ 2-3 κατά αποχές απορρίπτεται. 261 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 262. Αποσύρουμε, Πρόεδρε το αίτημα για ε, ψηφοφορία σε τμήματα, Επομένω μπορούμε να ψηφίσουμε ολόκληρο το κείμενο. Κύριο Φέρμα, ε, Πρόεδρε, εάν πρόκειται να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία 262, αν εγκριθεί, δηλαδή θα θέλαμε να μετακινηθεί στο σημείο 70β, 17β. Διακόσια... 62 λοιπόν, ολόκληρο το κείμενο, υπέρ. Κατά. Δύο ψήφοι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 263 υπέρ. Τρεις κατά. Υπόλοιποι αποχές ουδής. Τροπολογίες Επιτροπής Περιβάλλοντος μπορούμε να τι δούμε μαζί. Ωραία, όλες μαζί. 21 έω και 24 τη Επιτροπή Περιβάλλοντος υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτονται. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική 27 υπέρ. Κατά. Ουδής. Εγκρίνεται. Γυρίζουμε σελίδα. 270. Στροπολογία 270, υπέρ παρακαλώ. 4. Κατά. Οι υπόλοιποι. Αποχές. Απορρίπτεται. 271 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 273. Κατά. Είπαμε το υπέρ, όποιος θέλει το σηκώσει το χέρι του, στο κατά παρακαλώ, κατά για τη 273, σηκώστε το χέρι, ωραία, το. 274, υπέρ, Κατά. Απορρίπτεται. Αποχές πρέπει να ρωτήσουμε. 275 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 277 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 276 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 278 κατά παρακαλώ αποχές απορρίπτεται 279 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 280. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 283 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 287 υπέρ Μάλιστα. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. στην 287 ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 22 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. 289 υπέρ παρακαλώ. 6. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Δύο ψήφοι κατά αποχές. Ουδεμία. Εγκρίνεται. 295 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 29 υπέρ. Κατά. 2. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 302 302 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 30 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 314 υπέρ. 314 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 317 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 318 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 319 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 420 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 321 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 322 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 323 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 324 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 316 υπέρ. 6 κατά. αποχές απορρίπτεται. Κύριος Φέρμα. Άλλο ένα τεχνικό σχόλιο. Πιστεύουμε ότι το κείμενο της αρχικής παραγράφου της 34 αντιβαίνει με το συμβασμό 99. Αν ψηφίσουμε τη δική μας τροποποίηση και εγκριθεί δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αν ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο θα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί στην 34 λέμε ότι οι εγγύσεις θα πρέπει να καλύπτονται από την διαφορά κλπ με, τα, ε, με τις αιτήσει δαπάνες που έχουν εγγραφεί στον προπολογισμό. Στην 99 λέμε κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλάμε για την κορυφή, για την ε, οροφή. Η οροφή είναι πολύ διαφορετική από το περιθώριο, από τη διαφορά. Ε, αν ψηφιστεί η τροπολογία μας όμως αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Αυτή ήταν η συμβαστική 99 τώρα. Ο, μιλάς για το συμβασμό 99. Ωραία, η συμβαστική πρόταση 99 νομίζω θα ψηφιστεί, θα υπερψηφιστεί, οπότε θα αντικαταστήσει όλη την παράγραφο 34. Όχι, κάνω λαθός. Also, wenn das wirklich so sein sollte, dann... Όταν έρθει η ώρα θα το παληθεύσουμε πάντως. Κύριο Σεκχάουτ. Εν γέννη συμφωνώ με τον κύριο Πριν όμως τώρα δεν μπορώ να συμφωνήσω. Γιατί στις 34 μιλάμε για την κατάσταση όπως έχει τώρα, ενώ στις 39 εκφράζουμε τις επιθυμίες μας για το μέλλον. Άρα υπάρχει διαφορά. Και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την λογική του, αλλά ούτε και την τροπολογία. Καλώ λέει ο Πρόεδρο. Λοιπόν, ψηφίζουμε πώ είναι στον κατάλογο των ψηφοφοριών και στη συνέχεια θα δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τι άλλο ε, χρήζει ενδεχομένως νομοτεχνικής βελτίωσης, εφόσον, εφόσον χρήζει. 326. Τροπολογία 326. Υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε, παρακαλώ. Άλλο νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίες. 21 υπέρ, 26 κατά, καμία εποχή. Εντάξει, τα πρόλαβα τα είδα. 21 υπέρ, 26 κατά, 0 εποχές, 327 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 333. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 344 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπαριθμόν 3 τροπολογία της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 348 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 16α υπέρ. Κατά. Συμβαστική 34 υπέρ. Κατά. Αποχές μία. Εγκρίνεται. 357 τώρα. Κατά. Αποχές απορρίπτωτα. 358 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 359 υπέρ. Οχτώ. Κατά. Λοιπόν. Αποχές. Απορρίπτεται. 360. Κατά. Αποχές. το. 35 συμβαστική υπέρ. Κατά. Ένας αποχές εγκρίνεται. 376 υπέρ. Τέσσερις κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 389 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Και μετά δεύτερο. Υπέρ του υπαριθμών ένα τμήματος. Κατά του πρώτου τμήματος. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ε, σαφές το αποτέλεσμα. Σαφέστατο. 39 συμβαστική υπέρ κατά αποχές μία εγκρίνεται η 40 συμβαστική υπέρ κατά αποχές μία 405 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 406 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Συμβιβαστική 41 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερις στη Σίτρε τώρα. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Η 21 22, 23, 25 υπέρ, κατά, μάλλον 22 μέχρι 25. Αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 42 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τετρακόσια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 422 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 43 υπέρ κατά ψήφος ε, αποχές εγκρίνεται 431 υπέρ κατά αποχές απορρίπτω 432 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Επιτροπή Πολιτισμού Παριθμόν 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπαριθμόν 7 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αποχές. Απορρίπτεται. Επιτροπή των Γυναικών υπαριθμόν 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 44 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 435. Προσθήκη μόνο μιας φράσης όπως η Ρωμά. Υπέρ. Κατά. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά σε επαληθεύσουμε. Έτσι φαίνεται. Πέρασε τη ψηφοφορία. 25 υπέρ, 22 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Η Επιτροπή Γυναικών, υπαριθμών 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 444 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 445 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 447 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 448. Ζητώ συγγνώμη, λέει πρόεδρος. 449 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 και 9 πολιτισμού, 10 και 11, να μην τις ψηφίσουμε μαζί. Όχι, καλά. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απρίπτεται. 9 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική υπαριθμών 45 υπέρ κατά μια ψήφους αποχές εγκρίνεται της Επιτροπής Γεωργίας υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 461 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εγκρίνεται διορθώνει πρόεδρος 467 Όχι, προλαβαίνω και εγώ να το, δω, να το διορθώσω. 467 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, Επιτροπή Γεωργίας Παρθυπών λοιπόν 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμών 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται υπαριθμών 7 τη Επιτροπής Γεωργία μαζί με την 8 και την 9 μαζί. 7, 8, 9 γεωργιες υπερ υπέρ, αποχέ. αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 47α υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνονται. 47 β συμβιβαστική υπέρ. Επαληθεύουμε. Εντάξει, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ξεκινάει. Πρόκειται για την αρχή της αμοιβαιότητας. Πέρας προφορίας. 21 υπέρ, 25 κατά. Μία αποχή. Απορρίπτεται. Η 462 τώρα. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Καλώς. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ας απολυθεύσουμε. Για το πρώτο κομμάτι της 462 ηλεκτρονική απολύθευση. Πέρας. 25 υπέρ, 23 κατά, καμία αποχή. Ήταν οι αναλογίες κάπω κοντίνε. Δεύτερο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τετρακόσια το δεύτερο τμήμα πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ. Δεύτερο τμήμα της 490. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. 486 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. 488 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 489 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 491 και 492 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 493 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 494 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 495 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 496 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 497 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 498 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 499 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 500 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 501 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 502 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επιτροπή Γεωργίας από την 11 μέχρι και την 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Υπαριθμόν 3 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 505 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 48 υπέρ κατά 3 αποχές εγκρίνεται 510 δεύτερο τμήμα ως προσθήκη βέβαια 510 δεύτερο τμήμα ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 512 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 4 και οι 17 της Επιτροπής Γεωργίας παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται η 14 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά απορρίπτονται απορρίπτεται 48α συμβιβαστική υπέρ κατά μία ψήφος αποχές εγκρίνεται 515 ως προσθήκη υπέρ. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 515 ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Είναι προσθήκη. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. 516. Το αυτόν πρόκειται πάλι για προσθήκη δηλαδή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 520. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 της Επιτροπής Βιομηχανίας υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω να σηκώνω όλα τα χέρια τους. Βλέπω να κουράζεστε τώρα πια. Ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. 13 της Επιτροπής Βιομηχανίας, παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Ε, είναι σαφές. Να σηκώνει το χέρι λοιπόν το ΕΛΚ πότε πότε για να βλέπουμε ξεκάθαρα το αποτέλεσμα. 17 υπέρ, 31 κατά, απορρίπτωται. Η 10 και η 11 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50, συμβιβαστική 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 533 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 537 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 538 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13, 14, 15 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. 4 κατά. Όλοι οι υπόλοιποι αποχές. Απορρίψετε. Η συμβαστική υπαριθμών 51 υπέρ. Κατά. Λίγες ψήφοι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 548 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 549 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 550 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 551 υπέρ. Κατά. Περισσότερο λοιπόν. Κα... Αποχές. Απορρίπτεται. 552 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 553 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 554 υπέρ κατά Κατά παρακαλώ, κατά, κατά. Πρέπει λίγο να, να ξεκουνήσω το, ΕΚ. Κατά λοιπόν, αποχές απορρίπτεται 555 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος 3 έως και 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Συμβαστική 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 μέχρι και 19 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Χωριστά, λέει ο κύριος Φέρμου. Συγγνώμη, λέει. Πρόεδρος 16 υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 559 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 53 υπέρ. Κατά. Μία ψήφος. Αποχές. Εγκρίνεται. 571 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 573 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54α συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 584 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Κύριο Σάικερτ θα ήθελα να ψηφίσουμε την τροπολογία 595 των σοσιαλιστών γιατί υιοθετήσαμε τον συμβιβαστική πρόταση 55 που σου λέει ότι θέλουμε ε, ενέργεια, ενεργειακές υποδομές για όλα τα θέματα και αυτή η τροπολογία την άλλη μεριά των σοσιαλιστών τονίζει ότι η η χρηματοδότηση θα πρέπει να δίδεται κατά προτεραιότητα σε ε, ε, ε, project ανανεώσιμων ενεργειών, το οποίο σημαίνει ότι, δίνει μια προτεραιότητα. Από την άλλη λοιπόν λέμε ότι θέλουμε χρηματοδότηση για όλα τώρα. Αυτή η τροπολογία λέει ότι θα πρέπει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργεια να έχουν κατά το δυνατόν προτεραιότητα. Θα ήθελα να ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία. Ευχαριστώ. So leid es mir tut. Πριν όμως νομίζω ότι δεν είναι δυνατό. Δεν το επιτρέπουν οι κανόνες που έχουμε ορίσει εμείς οι ίδιοι. Όχι μόνο ο κανονισμός, αλλά οι κανόνες που ορίσαμε. Αν κοιτάξουμε λοιπόν τη συμβαστική τροπολογία, είναι σαφές το ποιες είναι οι προτεραιότητες μας και δεν μπορούμε να ορίσουμε νέα προτεραιότητα μέσα στην συμβαστική. Αυτό είναι το κείμενο. Όπως έχει, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ως προσθήκη. Παρακαλώ, πιστέψτε με, δεν επιτρέπεται. Εάν στο σημείο αυτό αποκλίνουμε από τον κατάλογο των ψηφοφοριών μας, θα τα κάνουμε σαλάτα σε άλλα σημεία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε τις ανώσιμες πηγές. Ε, όχι, κοιτάξτε να σας πω. Θα πρέπει να το αφήσουμε για την ψηφοφορία σε επίπεδο ολομέλειας στο θέμα αυτό. Με την τροπολογία αυτή που μπορούμε και πάλι να διατυπώσουμε όπως θέλουμε και να εισαχθεί το κείμενο εκεί που το θέλουμε. Αλλά όχι έτσι τώρα σε αυτή την ψηφοφορία και σε αυτό το σημείο καλύπτεται, έχει καλυφθεί, δεν μπορεί να μπει αυτό το, αυτή η πρόταση. Eichhardt. Δεν συμφωνώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πιστέψω, αλλά είναι μια πολιτική επιλογή κατά πόσον αποτελεί προτεραιότητα ή όχι. Εάν διαβάσετε τη συμβιβαστική πρόταση 55, δεν βάζουμε ε, κάποια προτεραιότητα. Λέμε ότι πολλά θα πρέπει να καλυφθούν από τις υποδομές ε, στην ενέργεια, ενώ εμείς θέλουμε να δοθεί προτεραιότητα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι προσθήκη στο 55. Θα ήθελα να σας πιστέψω, αλλά δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση δεν συμφωνώ μαζί σας και θα ήθελα να ε, ψηφίσουμε ξεχωριστές τις τροπολογίες. Also, δεν είμαι πεπισμένη ότι έχετε δίκιο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Βεβαίω μπορώ να το θέσω στην κρίση τη Επιτροπή. Θέλετε να γίνει ψηφοφορία νέου. Ναι Ένα λεπτό. Τώρα δεν ψηφίζουμε τις ε, προτεραιότητες για τις ανανεώσιμες πηγές. Αλλά το εάν επιτρέπεται να γίνει η σχετική προσαρμογή της τροπολογίας των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά μπορεί να αποφασίσει η Επιτροπή εάν θεωρεί ότι μπορούμε ή πρέπει μάλλον να ψηφίσουμε την δυνατότητα για ψηφοφορία της τροπολογίας αυτής. Ναι ή ου. Θέλουμε να γίνει ψηφοφορία για την τροπολογία αυτή, ναι ή όχι. Ποιο λέει το ναι, λοιπόν, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ναι, υπέρ τη εξαγωγής ψηφοφορία για την εν λόγω τροπολογία. Πέρας. Η πλειοψηφία στην Επιτροπή λέει όχι, δεν θα ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, ούτε καν ως πρόσθεκη. Και ο Μπάς και ο Γιώεραν το ξέρουν ότι η καρδιά μου χτυπάει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά θεωρώ ότι τεχνικά δεν είναι δυνατόν, δεν επιτρέπεται από τους κανόνες μας, επομένως σε επανέλθω το θέμα στην Ολομέλεια. Συμβαστική 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή των Μεταφορών, υπαριθμόν ένα υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 598 υπέρ κατά απορρίπτεται. Υπαριθμόν 2 τη Επιτροπής Μεταφορών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 583 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπαριθμόν 9 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 607 υπέρ κατά εγκρίνεται μάλλον, ναι. Συμβαστική 57 κατά αποχές εγκρίνεται. 618 ως προσθήκη based on a cost benefit analysis βάσει μιας ανάλυσης κόστους και ωφέλους. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επιτροπή των Μεταφορών. Τροπολογίε 12 έως και 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 619. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. και σα το λέω προκαταβαλικά τώρα για να μην ξαναρχίσει η ιστορία, η 627 θα έχει την ίδια τύχη με την 584 ε, ψηφίσαμε νωρίτερα, 584 ψηφίσαμε νωρίτερα, γι' αυτό λοιπόν προχωρούμε κατά άποχέ. απορρίπτεται 628 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Επιτροπή Μεταφορών, υπαριθμών 31. Α, όχι, έχει καταπέσει γιατί εγκρίθηκε 628. Καλώς. Συμβιβαστική 59. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 631 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 632 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 633 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 635 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60, συμβαστική 60 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ε, συμβαστική 61 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 652 ε, τροπολογία υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 συμβαστική υπέρ

κατά αποχές απορρίπτεται. Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, υπ. 19, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπερθυμών 64, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 της Περιφερειακής Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 694 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 695 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 65 υπέρ, κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 704 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 705 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επιτροπή των Γυναικών, υπαριθμών 15 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 709 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 721 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 724 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 723 τμήμα δεύτερο, το πρώτο έχει καλυφθεί, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περιφερειακή 15 και 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 744 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική υπαριθμών 70 τώρα. Και παρακαλώ κατευθείαν να περάσουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. SOD hat ein zu viel. Οι σοσιαλιστέ έχουν ε, μια ψήφο παραπάνω. Τώρα το ΕΛΚ έχει μια ψήφο παραπάνω, δύο μάλιστα. Jetzt stimmt's, wir schließen die Abstimmung. 30 dafür. 30 υπέρ, 15 κατά, δύο απόχέ. Η συμβαστική υπαριθμών 70 εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμό 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 756, πενήντα έξι υπέρ κατά αποχές απορρίψτε. 23 της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων υπέρ. Κατά. Αποχές. Απρίπτω. Συμβαστική. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. «758 υπέρ». Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 768 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 769 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 777 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και το ΕΛΚ το μετράω σαν ε, μία ομάδα γιατί είναι ο μόνος Ράιμαρ που σηκώσει το χέρι του Πες τους δικούς σου τέλος πάντων να σκόνουν και το χέρι. Απορρίπτεται λοιπόν. 778 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 779 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή Πολιτισμού 12 έως 24. Μπορούμε να τις δούμε όλες μαζί. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Επιτροπή Πολιτισμού 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 788 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πριν των πρασίνων. Επιτροπή των γυναικών με την τροπολογία παριθμών 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 807 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 808 υπέρ. Ταυτόσημη μάλλον. 809 διορθώνω λέει πρόεδρος. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 81. Πρέπει να ψηφίσουμε την 81. Συμβαστική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά έχουμε την 811 στο δεύτερο τμήμα μόνο, δεύτερο τμήμα της 811 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 814 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 815 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 819 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 818 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 816 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 817 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 820 υπέρ έχει αποσυρθεί εντάξει εντάξει αφού μου το είπατε εγκαίρως δεν υπάρχει πρόβλημα 865 υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται 82 συμβαστική 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επιτροπή Ανάπτυξης 1 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, απορρίπτονται συμβαστική 84 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 847 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 849 υπέρ Κατά. Η λυπή. Αποχές. Απορρίπτεται. Επιτροπή Ανάπτυξη Παριθμών 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, όχι, όχι, σοβαρά. Απορρίπτεται. 850 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ανάπτυξη. Από την 6 μέχρι και την 31. Υπέρ. Κατά. Κύριο Φέρμ. Χωρίς μικρόφωνο. Μέχρι την 30 λοιπόν. Ντέβε μέχρι 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Επιτροπή Ανάπτυξη Παριθμών 31, τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 851 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 852 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 853 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 854 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 855 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 856 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 της Επιτροπής Ανάπτυξης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 της Επιτροπής Ανάπτυξης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται διορθώνει ο Πρόεδρος. 842 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να υπαλληθεύσω αλλά μάλλον πάλι έχουμε το ίδιο φαινόμενο ότι δεν σηκώνετε το χέρι σας παρακαλώ λοιπόν 842 να υπαλληθεύσουμε Μάλλον θα έχει απορριφθεί. Πέρα προφορία 25 υπέρ 26 κατά. Καμιά εποχή. Εγκρίνεται. 857 υπέρ. Κατά. Αποχές. 858 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 859 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 860 υπέρ κατά εγκρίνεται εγκρίνεται με την αναλογία εγκρίνεται ναι, ναι. Ανάπτυξη 21-29. Πάντα με δυσκολεύεται. 21 με 28, άντε. 21 με 28. Κατά. Αποχές. 29 της ανάπτυξης. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 86 συμβαστική υπερθμόντα 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 868 υπέρ κατά απορρίπτεται 879 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 87 κατά αποχές εγκρίνεται 88 συμβαστική 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 878 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 882 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ, λέει πρόεδρος. Κατά... Ε, 90, συγγνώμη. Εγκρίνεται. ...844 τώρα... ...που μπορούμε να ψηφίσουμε ως, τελευταίο, ως προσθήκη στο τελευταίο του κομμάτι... ...844 ως προσθήκη στο τελευταίο κομμάτι... ...υπέρ... ...κατά... Εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε όμως. Πέρα προφορία 26 πέρα. 22 κατά. Εγκρίνεται. Ανάπτυξη παριθμών 7 αποχές απορρίπτεται. 885 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 συμβαστική 91 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 92 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 897 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεκαέξι επιτροπή Ανάπτυξης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 898 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 907 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 905 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 908 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 906 υπέρ Οχο. Μάλιστα. Πολύ καλά. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ αμέσως. Το ΕΛΚ έχει μια ψήφο παραπάνω. Κλείνω την ψηφοφορία. 22 υπέρ, 21 κατά, Τρεις αποχές. Χαίρομαι πολύ που το επαλήθευσα. 909. 909. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επιτροπή Μεταφορών υπαριθμών 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 101. Υπέρ. Κατά αποχές 8 ψήφι κατά. Ε, αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται στην επόμενη σελίδα, συμβαστική 94, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται συμβαστική 96 κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ 97 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 937 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 938 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ...951 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, συμβαστική υπαριθμών 100 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 953 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσω ηλεκτρονικά παρακαλώ Πάλι έχουμε μία ψήφο παραπανήση από το ΕΛΚ. Ας ε, επαληθεύσουμε λοιπόν. 24 υπέρ, 22 κατά. Αποχές δεν υπάρχουν, άρα καλά το κατάλαβα. 994 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ, 21 κατά. Αυτό που λέω εγώ είναι σωστό. Με κάποιε εξαιρέσει. Όταν με βοηθάει πάντω η ομάδα μου δεν υπάρχει πρόβλημα. Η αριστερή πάντως ε, πτέρυγα βλέπω πάντα να σηκώνει το χέρι με πολύ ε, ενεργητικότητα. Η δεξιά πτέρυγα κάπως πιο αδρανής. 970 παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 971 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 977 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 993 και λοιπές που είναι ταυτόσιμες υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 996 υπέρ. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ. Την 996. Πέρα στις προφορίες. Αχα. Απορρίπτεται. 105 συμβαστική. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Χίλια δεκαεφτά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1018 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107. την τελευταία εκδοχή του εισηγητού. Έτσι, την έχουμε λάβει όλοι. Δεν υπάρχει λόγο να συζητάμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάω στην 1028 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1029 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 1030. Υπέρ κατά. Σα τα λέω και ανάποδα. Πρώτα, πρώτα το κατά και μετά το υπέρ. Απορρίπτεται πάντω. Απορρίπτεται. 1031 υπέρ. Κατά. Καλά, δεν ανησυχούμε. Αποχές, απορρίπτεται 1032. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 108, άντε φτάσαμε. Ε, 108 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 110 αλφα υπέρ, κατά ηλεκτρονική επαλήθευση 110α. Ναι, είναι το σύστημα των ίδιων πόρων. Μπορούμε να το σώσουμε πάλι. Πέρας. 22 υπέρ, 26 κατά, χωρίς αποχές. Πάει και αυτό. Συμβαστική 111. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκατόν... 1080 ε, 1080 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την προφορική τροπολογία που έχουμε και στο τέλος ε, της παραγράφου αυτής. Το έχετε λάβει γραπτός. Το κείμενο υπέρ παρακαλώ. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Υπέρ της προφορικής τροπολογίας παρακαλώ για την παράγραφο 118 το έχετε λάβει ήδη το κείμενο. Πέρας της ψηφοφορίας. 19 υπέρ 29 κατά, οχιές δεν υπάρχουν. 1084 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1089. 1089 υπέρ. Κατά. ποιες απορρίπτεται. 1090 υπέρ. Κατά. ποιες απορρίπτεται. 1092 υπέρ. Κατά. ποιες απορρίπτεται. Συμβαστική 114 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα λίγο πολύ κλείσαμε την έκθεση και περνάμε σε θεολογικές σκέψεις και θεολογικές αναφορές και έτσι θα πάρουμε και μια μεγάλη ανάσα για να δούμε μπορούμε να τα πάρουμε όλα μαζί on block ωραία ευχαριστώ πολύ Παριθμόν 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επτά. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επτά. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εννέα υπέρ. Εννέα κατά. Όχι. Απορρίπτεται. Δεν υπάρχει λόγος να επαληθεύσουμε. Δέκα υπέρ. Κατά. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Έντεκα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Ας το επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε. Πέρασε προφορές. Αχα. 23 υπέρ, 25 κατά. Μάλιστα. Άρα θα ελέγχουμε από εδώ και μπρος. 12. Τροπολογία 12 υπέρ. Επαληθεύουμε. Επαληθεύουμε. Βλέπω ότι είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πέρες φοφορίες. 23 υπέρ, 25 κατά. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική παριθμόν 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τιολογική σκέψη ΔΕΛΤΑ τροπολογία 26 υπέρ. Νομίζω θα έχουμε τις ίδιες αναλογίες, αλλά θα το ηλεκτρονικά παρακαλώ την 26. Πέρας της προφορίες 25 υπέρ 23 κατά το ανάποδο αποτέλεσμα, το αντίστροφο αποτέλεσμα που περιμέναμε, δεν είναι δυνατόν να το προβλέψουμε λοιπόν. Η, η τροπολογία 27 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε την 32. Ας επαληθεύσουμε την 32. Πέρασε. 23 υπέρ, 25 κατά αυτή τη φορά. Απορρίπτεται δυστυχώς. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επιτροπή Γυναικών Β υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3α 3, α 3α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σαράντα οκτώ, τροπολογία σαράντα οκτώ. Καταπίπτει. Τι λέει. Α, καταπίπτει μάλιστα. Σαράντα εννέα λοιπόν. Σαράντα εννέα υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αγαπητοί μου φίλοι, τελευταία σειρά. πια. 53. Τροπολογία υπέρ 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Μάλιστα, καταπίπτει η πόρτα σα. Ε. Λόγω της 58. Και η 70 καταπίπτει. Επιτροπή των Γυναικών, τροπολογία C, Γ. Επιτροπή Γυναικών, τροπολογία C, Γ. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτω. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η Επιτροπή περί Ανάπτυξης A μέχρι D, Α έως και Δέλτα, χωρίς αντίρρηση. Ευχαριστώ. Υπέρ. Τρεις. Κατά. Η λυπή. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Στην έκθεση, στο σύνολό της, όπως τροποποιήσαμε με τις τροπολογίες που ψηφίσαμε όλοι μαζί. Παρακαλώ. Ηλεκτρονική λοιπόν ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε αρκετά μέλη από τους Ένας από το ΕΛΚΑ και ένας από τους σοσιαλιστές περισσεύουν. Ακόμη από τους σοσιαλιστές. Εντάξει. Τώρα είμαστε εντάξει με τα νούμερα. Πέρα στις ψηφοφορίες. 39 υπέρ, 5 κατά, 4 εποχές. Συγχαρητήρια κύριε Καγεύου. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την αντοχή, την αιμονή και την επιμονή σας, όχι μόνο στην ψηφοφορία, αλλά και για την πολύ, πολύ, πολύ καλή δουλειά που κάνατε. Άντε και καλή ξεκούραση τώρα.